σκόπιμο να την υποστηρίξετε μέσα στα πλαίσια της αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κάτσμαρεκ. Γραπτή δήλωση 0101 του 2012 για την μέρα, την εισαγωγή τη μέρα του, της μέρας του παραδοσιακού παγωτού. die von Ντεκάστρο, Μέλτσερ, Ορτής Βιλέγια και Στάντλερ. η δήλωση συγκέντρωσε την πλειοψηφία των μελών του Κοινοβουλίου και βάσει του άρθρου 123 του κανονισμού θα ε, διαβιβαστεί στους ε, παραλήπτες και θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά ως εγκριθέν κείμενο της συνεδρίασης. Επ' αυτού ο κύριος Σιλβέστρη ζητεί το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η μέρα αυτή θα γιορταστεί σε όλη την Ευρώπη στις 24 Σεπτεμβρίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που υπέβαλαν μαζί τη δήλωση για τους συναδέλφους Κοτέ και Σταγκαντζάν που υποστήριξαν τη δοκιμή παραδοσιακού ε, παγωτού στο Κοινοβούλιο, επιτρέποντα σε όλου πέρα από το να πάρουν την υπογραφή του να δοκιμάσουν και το παραδοσιακό παγωτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του παραγωγού που ήρθαν μέχρι το Στρασβούργο για να προσφέρουν τα παγωτά του. Η υποστήριξη του παραδοσιακού παγωτού σημαίνει το να προωθήσει κανεί ε, την αγνότητα του παγωτού και τα καλύτερα θρεπτικά συστατικά. Το παραδοσιακό παγωτό παράγεται ε, στον τόπο και υποστηρίζει τις ε, τοπικές γαλακτοκομικές μονάδες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους υπέγραψαν. So. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, περνούμε στις ψηφοφορίες τώρα. Έκθεση Τάιν. Ε, πρόκειται για το πρωτόκολλο για τον Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η κυρία Τάιν έχει το λόγο, η συγγήτρια. Αξιότιμη